Uh, Νομίζω ότι μπήκαν στην αίθουσα όσοι ήθελαν να μπουν. Κύριο Ζεύκα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εξετάζουμε τρεις εκθέσεις ε, για τις οποίες είμαι εισηγητής. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση που αφορά τις διασυνοριακές πτυχές που αφορούν οι οθεσίες παιδιών. Αυτό οφείλεται σε κάποια προβλήματα υγείας που είχα ήμουν στο νοσοκομείο, αλλά ελπίζω ότι από εδώ και πέρα θα προχωρήσουμε με ταχύτητα και θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες και να προετοιμάσω την τελική έκδοση αυτής της έκθεσης πριν το τέλος του 2016. Το σχέδιο έκθεσης αυτό εστάλει πριν από δύο εβδομάδες και έχει δύο τμήματα. Το πρώτο μέρος της έκθεσης ακολουθεί τέσσερις προσανατολισμούς τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές. Κατά την άποψή μου με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνουμε τα σημαντικότερα σημεία τα οποία είχαμε συζητήσει εδώ μεταξύ μας αλλά και κατά την ακρόαση που οργανώσαμε στο τέλος του 2015. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση και μας βοήθησε πολύ έτσι ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το θέμα αυτό. Καταρχήν, τα ελάχιστα πρότυπα. Αυτά τα ελάχιστα πρότυπα θα πρέπει να διέπουν όλες τις περιπτώσεις υιοθεσία, ιδιαίτερα όμως όταν πρόκειται για διασυνοριακή υιοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κοινά ελάχιστα πρότυπα. Όλοι συμφωνούμε ότι το συμφέρον του παιδιού είναι καθοριστικό και στο κέντρο της διαδικασίας. Το συμφέρον του παιδιού λοιπόν πρέπει να είναι η καρδιά της διαδικασίας και κανένα σύστημα νομικό σε καμία χώρα δεν θα πρέπει να θεωρεί το παιδί σαν ιδιοκτησία ενός ενήλικα ή ενός ε, ζευγαριού. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε με αυτήν την ε, κατευθυντήρια γραμμή, οδηγούμαστε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας σε κάθε περίπτωση τα πιο κοντινά πρόσωπα του παιδιού σε όποια χώρα και αν διαμένουν. Και κατά τη διάρκεια της ακρόασης είδαμε ότι όλα τα παιδιά, ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους, εάν βεβαίως συμφωνούν και οι βιολογικοί γονείς. Κατόπιν, στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, αναφερόμαστε στην έκθεση της Χάγης του 1993, που αφορά την προστασία του παιδιού, τη συνεργασία όσον αφορά την ε, διεθνή υιοθεσία, και παρόλο που λειτουργεί με πολύ ικανοποιητικό τρόπο αυτή η σύμβαση της Χάγης για την υιοθεσία των παιδιών τα οποία ζουν, κατοικούν σε μια διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία βρίσκονται οι γονείς, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές παρόλα αυτά όσον αφορά κυρίως την προσέγγιση όσον αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων που ουσιαστικά επιβάλλει η Σύμβαση της Χάγης. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχουν κάποιες διαφορές, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσπαθήσουμε να τις εξισορροπήσουμε, να τις περιορίσουμε ή να τις εξαλείψουμε, αν αυτό είναι δυνατόν. Υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες που αφορούν τα πιστοποιητικά υιοθεσίας. και αυτές οι δυσκολίες και τα προβλήματα προκύπτουν παρόλο που η Σύμβαση θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει αυτόματη αναγνώριση της υιοθεσία από όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν λειτουργεί στο σημείο αυτό ικανοποιητικά η Σύμβαση παρόλο που διοικητικές διαδικασίες υπάρχουν, παρόλο που τα κράτη-μέλη που έχουν ε, κυρώσει τη σύμβαση έχουν δεχτεί όλες τις, τις διατάξεις. Βλέπουμε όμως ότι πρόκειται για μια διασυνοριακή συνεργασία η οποία περιέχει προβλήματα, συνεργασία μεταξύ των δικαιοδοτικών οργάνων, μεταξύ των θεσμικών οργάνων των ε, κρατών μελών. Πρόκειται για τα θεσμικά όργανα αυτά, τα οποία δικαιωματικά μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες υιοθεσία. Ένα άλλο θέμα είναι η διασυνοριακή αυτή αναγνώριση των πιστοποιητικών υιοθεσία και των διαδικασιών υιοθεσία των διαφορετικών χωρών. Είναι καθοριστικό το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο διασφαλίζει την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τμήμα αυτό της έκθεσης έχει σχέση και με το παράρτημα. Και έρχομαι στο πιο σημαντικό θέμα αυτής της έκθεσης. Προτείνω λύσεις, ευρωπαϊκές λύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την υιοθεσία που λαμβάνει η χώρα σε μία χώρα σε κάποιες άλλες χώρες. Τώρα, θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω και τα σημεία τα οποία δεν καλύπτει η έκθεσή μου. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αλλάξω τον κανονισμό. Δεν επιθυμώ να τροποποιήσω την νομοθεσία, της διατάξεις που αφορούν την υιοθεσία στα κράτη-μέλη. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε εδώ να επέμβουμε στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Δεν ζητούμε από τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν νομικούς δεσμούς μεταξύ του παιδιού και των βιολογικών γονέων. Εάν και εφόσον η εθνική νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Το σχέδιο έκθεσης μου ζητάει την αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών υιοθεσία χωρίς να υπάρξει απολύτως καμία επιπλέον διαδικασία. Αυτό μπορεί να συμβεί υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, εάν ένα κράτος μέλος διαθέτει μία αρμοδιότητα που να του επιτρέπει να δώσει ένα τέτοιο πιστοποιητικό και δεύτερον, εάν μια τέτοια απόφαση δεν αντιτίθεται στην ομοθεσία δεν αντιβαίνει στην νομοθεσία του κράτους μέλους που πρέπει να αναγνωρίσει την διαδικασία της υιοθεσία. Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένε ρήτρε οι οποίες ε, εφαρμόζονται εάν ένα διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό υιοθεσία απορρίπτει το αίτημα. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό αναγνωρίζεται από το κανονισμό Βρυξέλλες 2 και Ρώμη 3. Ο κανονισμός αυτός, συγγνώμη, η έκθεση αυτή προτείνει επίσης και την ε, ύπαρξη ενός πιστοποιητικού για την ε, μετακίνηση των ε, γονέων με το παιδί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Πρόκειται για μια απλοποίηση όλων των διαδικασιών που δυσκολεύουν σήμερα τη ζωή των γονέων. Γιατί η διαδικασία σήμερα είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Προσθέτω επίσης και όλα τα έντυπα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν για να υπάρξει αναγνώριση της διαδικασίας υιοθεσία. Περιγράφω τις περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει απόρριψη ε, ε ενός τέτοιου αιτήματο και τις πιθανές προσφυγές. Περιγράφω δηλαδή όλες τις δυσκολίες και περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι το σχέδιο κανονισμού που υποβάλλεται στο παράρτημα βασίζεται επίσης στην ανάλυση που έχει γίνει από αυτήν την ομάδα αξιολόγησης της προστιθέμενης ε, ευρωπαϊκής αξίας και φυσικά λαμβάνουμε υπόψη μας ε, ε, αυτήν την γνωμοδότηση. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε πως σε όλες τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διαδικασίες υιοθεσία είναι διαφορετικές. Γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι μετακινούνται, μετακομίζουν από τη μία χώρα στην άλλη, αντιμετωπίζουν πλήθος δυσκολιών και προβλημάτων. Και όσον αφορά κάποιες ε, χώρες, πολλές φορές τους κατηγορούν ότι έχουν ε, πάρει το παιδί από τους βιολογικούς γονείς. Σε άλλες ε, χώρες οι διαδικασίες υιοθεσίας μπορούν να κρατήσουν χρόνια και είμαι πεπισμένος ότι η απόφασή μας, η δράση μας θα διευκολύνουν και θα επιλύσουν πολλά από αυτά τα προβλήματα. Θα διευκολύνουν τους ε, γονείς που θέλουν να υιοθετήσουν. Όσον αφορά τις τροπολογίες, σας προτείνω την προθεσμία υποβολής 30 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Έφτασε η ώρα 10 όμως και είναι η ώρα για τις ψηφοφορίες. Σας προτείνω να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για τις ψηφοφορίες και να συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα μετά την ψηφοφορία. Γιατί και έχουν έρθει οι συνάδελφοι για την ψηφοφορία. Please make sure you have your voting cards. Σας παρακαλώ πολύ να εξασφαλίσετε πως έχετε τις ε, κάρτες σας.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 Ο εισηγητή σα μα δώσει λίγο, μάλλον ο εισηγητής έχει φύγει από την αίθουσα. Περιμένουμε τον κύριο Καβατά για λίγα δευτερόλεπτα, άρα λοιπόν ας κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Okay. Uh, article 3, paragraph 1. Λοιπόν, 3, 1, ε, α, υπέρ. Against. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64α υπέρ Against. Κατά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Ο κύριος Ζεύκα είναι υπέρ. 11-11. Απορρίπτεται λοιπόν. Ηλεκτρονικά λοιπόν θα έχουμε και τη σχέδιο έκθεση, θα το ψηφίσουμε ολόκληρη την έκθεση. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Εγκρίνεται. Έχουμε μετά το ψήφισμα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Εγκρίνεται. Σχέδιο έκθεσης ολόκληρο. Adopted. Εγκρίνεται λοιπόν. Και το σχέδιο ψηφίσματος ξεκινάει ψηφοφορία. Επίσης εγκρίνεται. Θα ήθελα να σας συγχαρώ λοιπόν, κύριε Σίτα. Ο οποίος δέχεται τα συγχαρητήρια και σας ευχαριστεί. That is the end of the vote. And we may... Τελείωσαν οι ψηφοφορίες, μπορούμε τώρα να περάσουμε με το σημείο 24. Θα ήθελα τώρα... Sorry? Uh, okay, we'll go back to that one. Uh, do we have Mrs. Ruth Cabeza? Καταρχήν θα ήθελα να δω αν έχουμε τη συνάδελφο Ρουκαπέτσα στην αίθουσα. So, uh, madam, uh, we have time now. Κυρία μου, έχουμε μέχρι τις 10 και μισή. Αλλά χρειαζόμαστε και τις ερωτήσεις των μελών να ακούσουμε. Οπότε Έχετε 18 λεπτά στη διάθεσή σας για να γίνουν όλα αυτά. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Mr. Chairman, members. Uh, Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτήν την ενδιάμεση αξιολόγηση για το θέμα της διασυνοριακής ε, πτυχής ε, των, ε, αναγνώρισης των ε, υιοθεσιών. Είναι το κείμενο της κυρίας Ρούθ Καμπέσα. Το έχει προετοιμάσει λοιπόν η γενική μας διεύθυνση και ήθελα να σας πω ποιος είναι ο στόχος. Είναι να στηρίξουμε τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζοντας προς το πολύ τα νομικά στοιχεία που τεκμηριώνουν πως αξίζει να λάβουμε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ κάνουμε και μια ποιοτική ανάλυση αλλά και μια ποσοτική ανάλυση της προστιθέμενης εξία του να κάνουμε τέτοιου είδους νομοθετικές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν περάσουμε λοιπόν στην πέμπτη διαφάνεια για να σας παρουσιάσουμε το τι διακυβεύεται, λοιπόν, οι διασυνοριακές υιοθεσίες ρυθμίζονται σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών από τη Σύμβαση της ΧΑΙΣ του 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία για τις διασυνοριακές υιοθεσίες. Στο άρθρο 23 συμπεριλαμβάνει την αυτό αυτόματη αναγνώριση των διαταγών υιοθεσία. Αλλά το πεδίο εφαρμογή της σύμβαση είναι περιορισμένο. Καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις όπου και το υιοθετημένο παιδί και οι υιοθετούντε γονεί διαμένουν σε δύο διαφορετικά κράτη-μέλη. Στην περίπτωση που διαμένουν στο ίδιο κράτος μέλος δεν καλύπτεται από τη Σύμβαση της Χάγης, αντίθετα υπόκεινται στο εθνικό δίκαιο. Αυτό βεβαίω δημιουργεί ένα νομικό κενό και υπάρχει μια δικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των νομικών ε, επιπτώσεων που έχει η Σύμβαση της Χάγης με την εθνική νομοθεσία όταν υπάρχει κάποιο στοιχείο ολοδοπό, για παράδειγμα διπλή υπηκότητα του γονιού που υιοθετεί. Άρα λοιπόν έχουμε αυτόματη αναγνώριση με τη Σύμβαση ε, Χάγης, ενώ οι εθνικές υιοθεσίες δεν αναγνωρίζονται αυτόματα από κάποιο άλλο κράτος μέλος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό έχει αρνητική επίπτωση κυρίως για οικογένειες οι οποίες ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ούτε για το παιδί, ούτε για το γονέα πως η, το καθεστώς υιοθεσία και οι νομικές επιπτώσεις θα αναγνωριστούν εάν η οικογένεια αποφασίσει να ζήσει σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό βεβαίως επιφέρει και κάποιο κόστος. Αν κοιτάξετε στο, στη διαφάνεια 4 θα δείτε πως το κόστος που απορρέει από την έλλειψη ε, κοινοτικών κανόνων στην αναγνώριση αυτών των αποφάσεων υιοθεσία και εδώ κάνω ένα χαμηλό υπολογισμό, είναι περίπου 1,65 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και αυτό ε, καλύπτει μόνο τα δικαστικά έξοδα. Και αυτή η έκθεση αναλύοντας το κόστος αλλά και τα ωφέλη από την νομοθεσία εμείς προκρίνουμε να δημιουργηθεί ένα δεσμευτικό μέσο ε, για τις υιοθεσίε και την αναγνώριση των ε, σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 81 της ε, συνθήκης με αυτόματη αναγνώριση των εθνικών αποφάσεων υιοθεσία που μας φέρνει στη διαφάνεια που είναι η εναλλακτική 2, option 2, που είναι ένας δεσμευτικός κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων υιοθεσία. Με στόχο εδώ να δώσουμε την απαραίτητη βεβαιότητα για το καθεστώς των υιοθετημένων παιδιών και δεν έχει στόχο να ε, παρέμβει στο εθνικό δίκαιο που διέπει τις υιοθεσίες. Δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν την ελευθερία να νομοθετήσουν όσους θεωρούν σωστό για ε, το ποια παιδιά θα πρέπει να δίδονται σε ε, υιοθεσία, για τον τρόπο που θα γίνεται η υιοθεσία, για τον τρόπο που θα ε, επιλέγονται οι γονείς, αλλά το μόνο που ρυθμίζει είναι η αναγνώριση των αποφάσεων υιοθεσία από τα εθνικά δικαστήρια. Αυτά ήθελα να πω. First of all, let me thank you very much. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εμένα και το συνάδελφο και τους συναδέλφους μάλιστα να προετοιμάσουμε αυτό το, αυτή τη μελέτη και είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ. Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να απαντήσω είναι η εξής. Γιατί χρειάζεται να νομοθετήσουμε. Οι περισσότεροι δικηγόροι θεωρούν πως το σχέδιο που ε, προετοίμασε η συγγήτρια ήδη υπάρχει, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία διάταξη που να εξασφαλίζει το καθεστώς των παιδιών που θετήθηκαν υπό τους εθνικούς νόμους ή από τα δικαστήρια ενός κράτους μέλους σε όλη την Ευρώπη ή τουλάχιστον σε όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος μέλος το οποίο εξετάσαμε στα πλαίσια της έρευνάς μας έχει διατάξει εθνικές για την αναγνώριση των των αλλοδαπών αποφάσεων υιοθεσία, αλλά κάθε κράτο μέλο έχει διαφορετική διαδικασία. Άλλε είναι πιο απλέ, άλλε όχι. Και από τη στιγμή που έχει δοθεί αναγνώριση, ε, εφαρμόζεται βέβαια μόνο στο οικείο κράτο μέλο. Και ακόμα περισσότερο όταν η σχέση γονέα-παιδιού αναγνωρίζεται, αυτό δεν σημαίνει πω αυτομάτω το παιδί είναι σε. Ε, σε ίση μοίρα με το παιδί του παιδιού που έχει οθετηθεί σύμφωνα με τον νόμο του ε, άλλου κρατούς μέλους. Για παράδειγμα, ε, έχουμε κάποιες ε, αναγνωρισμένες αποφάσεις αλλοδαπής ε, που επιτρέπουν πιο εύκολες διαδικασίες απόκτησης της ηθαγένης με συγχωρείτε, της υπηκότητας του γονέα που υιοθετεί. Αυτό που μας απασχολεί είναι ποια είναι τα πιο ευάλωτα παιδιά και αυτά και τα παιδιά που είναι ευάλωτα είναι ε, τα παιδιά τα οποία υιοθετούνται από οικογένειες οι οποίες μετακινούνται πολύ, όπου ε, δεν έχουν την ίδια υπηκότητα ε, με τους γονείς τους και όπου βεβαίως το ζευγάρι μπορεί να έχει και διαφορετικές υπηκότητες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μπερδευόμαστε με τις διασυνοριακές υιοθεσίες με αυτούς που γίνονται μέσα στο ίδιο το κράτος μέλος. Υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία και λυπάμαι που τρέχω, αλλά έχουμε την περίπτωση μιας διασυνορικής υιοθεσίας στο οποίο μπλέκονται δύο κράτη. Σύμφωνα λοιπόν με την σύμβαση του 1993 εκεί που ε, διαμένει συνήθω το παιδί είναι το κράτο προέλευση. Και εκεί που συνήθω διαμένουν οι γονεί είναι το κράτο υποδοχή. Μόνο το κράτο προέλευση ή το κράτο υποδοχή έχουν τη δυνατότητα να διατάξουν η οθεσία για ένα παιδί. Και όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεχτεί αυτόν τον περιορισμό στην, ε, στην δυνατότητα τη ε, διαταγή υιοθεσία στα πλαίσια του εθνικού δικαίου. Και τι λέει η Σύμβαση τη Χάγη, πως είναι το κράτος που ε, το κράτος προέλευσης που έχει τη δικαιοδοσία για να δικάσει το κατά πόσο ένα παιδί θα πρέπει να δοθεί σε υιοθεσία και αν είναι κατάλληλο η υιοθεσία διασυνοριακά. Η πρόταση δική μας βασίζεται λοιπόν σε αυτές τις αρχές και εμείς προτείνουμε το κράτος μέλος να έχει δικαιοδοσία για ε, διαταγή υιοθεσίας που να περιορίζεται σε περιπτώσεις που το παιδί είτε διαμένει σε εκείνο το κράτος μέλος είτε δεν διαμένει ε, είτε δεν διαμένει συνήθως σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Και στην πρότασή μας, όταν το παιδί και ο γονέας έχουν συνήθει διαμονή στο ίδιο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα πρέπει να είναι αυτό το κράτος μέλος το οποίο θα έχει τη δικαιοδοσία να ε, δώσει μια διαταγή υιοθεσία για το συγκεκριμένο παιδί. Στο άρθρο 24 της Σύμβασης του 1993 λέγεται πως η αναγνώριση μιας υιοθεσία μπορεί να μην γίνει από συμβαλόμενο κράτος, να μην δοθεί από συμβαλόμενο κράτος, μόνο αν η υιοθεσία είναι προδειλα ε, ε, σε αντίφαση με ε, τις δικές του διατάξεις, ε, πρόδειλα εναντίον του συμφέροντος του παιδιού και η αναγνώριση που θα δεχτούμε εμείς θα πρέπει να ακολουθεί αυτές τις, ε, αυτή τη διατύπωση που αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη-μέλη ως βάση για την απόρριψη μιας καταλήλως αποδεδειγμένης και τεκμηριωμένης απόφασης υιοθεσίας. Αυτό μας δίνει ένα μεγαλύτερο πεδίο για να αρνηθούμε να αναγνωρίσουμε μια διαταγή υιοθεσία και αυτό το σημείο θα πρέπει να το εξετάσουμε γιατί πιστεύω ότι στο θέμα τη αναγνώριση, μια μόλι συσταθεί σα οικογένεια αυτό που έχουμε στο άρθρο 8 θα πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού το οποίο θα πριτανεύσει και όχι η δημόσια πολιτική που ακολουθεί το ε, κράτος μέλος που ε, σκοπεύει να ε, απορρίψει αυτή τη διαταγή υιοθεσίας. Δεν θέλω να ε, χρησιμοποιήσω και άλλο χρόνο. Βρίσκονται όλα στη μελέτη, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πως οι προτάσεις μας και οι προτάσεις δικές σας είναι στα είναι ε, σίγουρα στα πλαίσια του άρθρου 67 και 81 και νομίζω πως η εκτεταμένη νομοθεσία που υπάρχει δεν είναι πολύ διαφορετική από ε, τις περιπτώσεις που έχουμε αναγνώριση αποφάσεων στις αστικές υποθέσεις και για την ευθύνη του γονέα δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να ε, εξυπηρετεί τους στόχους ε, αυτών των υιοθεσιών ε, και δεν νομίζω ότι μπορούμε εδώ να καταφέρουμε κάτι εάν η νομοθεσία που θα εισάγουμε δεν θα ισχύσει όλα τα κράτη-μέλη. Στη μελέτη μας αυτή λέμε πως προτείνουμε να υπάρξει νομοθεσία, ίσως ένα λιγότερο παρεμβατικό μέσο, αλλά είμαστε σίγουρα υπέρ της σκέψης πως οι μη δεσμευτικέ κατευθυντήριε γραμμέ ε, ε, και μια οδηγία δεν θα καταφέρουν να πετύχουν το στόχο μα, που είναι ένα απλό και αυτόματο τρόπο για να διχορηγείται η αναγνώριση. Και ότι μια οδηγία κυρίω θα μπέρδευε περισσότερο αυτό το ad hoc σύστημα αναγνωρίσεων που ήδη υπάρχει. Δεύτερον, θεωρούμε πω οποιοδήποτε άλλο τρόπο ε, για την αναγνώριση υιοθεσιών θα πρέπει να ξεκαθαρίζει πω είναι διαφορετικό το πλαίσιο για τι εθνικέ υιοθεσίε ε, νομίζω αυτό το νομικό θέμα το έχω ήδη καταλήλως εξηγήσει και συστήνουμε πως ε, μετά από μια εθνική διαταγή οθεσίας θα μπορούσαν οι γονείς να ζητούν ένα πιστοποιητικό από τις κεντρικές αρχές του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει τη διαταγή οθεσίας για να αποδεικνύεται η αυθεντικότητα αυτής της διαταγής και πως όλα ε, τα μέλη του άρθρου 6 να έχουν εξασφαλίσει τα δικαιώματά του στα πλαίσια τη διαδικασία υιοθεσία. Επίση, συστήνουμε, εφόσον έχει πιστοποιηθεί μια υιοθεσία, να είναι υποχρεωτικό όλα τα κράτη-μέλη να αναγνωρίζουν αυτή την υιοθεσία μέσω ε, νόμου, εάν ε, σαν να είχε γίνει αυτή η οθεσία στα πλαίσια του εθνικού δικαίου αυτών των κρατών μελών. Δεν θεωρούμε από το, ότι η προσέγγιση που ισχύει σήμερα ε, είναι επιτυχημένη ε, και θέλουμε η νέα νομοθεσία να βασιστεί στις επιτυχίες της Σύμβαση του 1993 και να πάει λίγο πιο κάτω. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα απόρριψη αναγνώρισης αλλά μόνο υπό περιορισμένες συνθήκε στα πλαίσια του άρθρου 24 τη Σύμβαση τη Χάγη. Για την προστιθέμενη αξία που θα προσφέρει κάτι τέτοιο, θα πω μόνο και θα προσθέσω στα όσα είπε η συνάδελφος πως οι διατάξεις στις, ε, στη μελέτη μας θα δώσουν ε, νομική βεβαιότητα στο καθεστώς του παιδιού, θα ησυχάσουν οι γονείς ότι χρειάζεται να περάσουν μόνο μία νομική διαδικασία, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται η υιοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ισότητα μεταχείριση στι οικογένειε που μετακινούνται και που έχουν υιοθετημένα παιδιά, έτσι ώστε τα δικαιώματα του υιοθετημένου παιδιού να είναι τα ίδια με τα δικαιώματα των παιδιών που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας του κράτου μέλου που αναγνωρίζει και επίσης μια ε, οικονομικά ωφέλη για την οικογένεια γιατί δεν θα χρειάζεται να λάβουν νομική συνδρομή είτε ε, να περάσουν από δικαστική διαδικασία σε κάθε κράτος όπου θα χρειάζεται αναγνώριση. Αλλά επίσης και για το κράτος το οποίο επιδιώκεται αναγνώριση το κόστος της διεκπαιρέωσης, της καταχώρησης της δικαστικής διαδικασίας για την αναγνώριση. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ για τις εισηγήσεις αυτές. Σχόλια από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους και ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Και η συνάδελφος Βιρζινή Χοζιέχ ε, έχει κάνει αυτή την πρόταση, ε, την οποία σας διαβάζω στα γαλλικά. Κύριε Ροζιέ, θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης και συμφωνεί με τον βασικό στόχο. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αυτόματη αναγνώριση σε ένα κράτος μέλος της απόφασης περί η οποία λαμβάνεται σε άλλο κράτος μέλος. Αυτά είναι στα σημεία 8 και 17. Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι απαραίτητη για να προστατεύονται καλύτερα τα παιδιά καταρχήν, αλλά και για να υπάρχει εγγύηση ασφάλειας δικαίου και προστασία των δικαιωμάτων των γονέων. Επιπλέον, αυτό θα ενισχύσει το συνέστημα του ανήκειν και της ευρωπαϊκής ηθαγένειας και την ε, καθημερινή ασφάλεια των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ντοχοζιέ τονίζει επίσης ότι συμφωνεί με πολλά από τα σημεία στην έκθεση, στην έκθεση ε, του εισηγητού, όπως είπε ο κ. για το συμφέρον του παιδιού που πρέπει να προέχει και το κύριο συμφέρον του παιδιού και το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι το κύριο κριτήριο βάσει του οποίου θα λαμβάνεται η αδίποτε απόφαση σε σχέση με την υιοθεσία. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, να διασφαλίζουν την ε, τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών και να φροντίζουν οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση την ε, ηλικία και την οριμότητα του παιδιού. Τώρα, κάποιες διατυπώσεις, σύμφωνα με την κυρία Ντροζιέρ, πρέπει να ε, τις επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο στο σημείο Β και Γ συγκεκριμένα, σε κάποιο σημείο του παραρτήματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, πολύ σημαντική δουλειά που κάνατε. Η κυρία Ντροζιέρ προσβλέπει στη συνεργασία με τον κύριο Σβέφκα και τους άλλους και συζητητές. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την εις βάθος ε, ε, ανάλυση του συναδέλφου Σβίφκα. Θα επανέλθω σε ένα λεπτό σε αυτήν και να ευχαριστήσω και τις εμπειρογνώμονες που ε, μόλις πήραν το λόγο γιατί υπάρχει ε, όντως ανάγκη να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κείμενο ομοιόμορφο ε, για αυτή την υπόθεση, την υιοθεσία παιδιών, την προστασία των παιδιών αλλά και την προστασία των γονιών αυτό το οποίο εκτιμώ όλος ιδιαίτερας είναι ότι επιτέλους βγαίνουμε από την αμφισημία την οποία είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο για πολλά χρόνια για αυτό το θέμα. Θυμηθείτε τα παιδιά της Ρουμανίας το 2005 και άλλες σχετικές εκθέσεις διαδοχικές όπου το Κοινοβούλιο ήταν διχασμένο, διαιρεμένο και δεν υπήρχε και βάση για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε. Να πω κάτι κάπως ε, βίο. Εδώ και αρκετές δεκαετίες ρυθμίσαμε το πρόβλημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ε, εμπορευμάτων και των υπηρεσιών. Αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν πια, αλλά μας χρειάστηκαν στην ουσία πέντε δεκαετίες για να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και, κυρίως, ιδίως τα παιδιά για την ελεύθερη κυκλοφορία και τους γονείς που τα βοηθούν, που τα υιοθετούν και που πολλές φορές εκτίθεται σε διώξεις αλλά και σε κόστος οικονομικό και πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δουλειά γιατί έπρεπε να δώσουμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτή την ένωση που αντιμετωπίζει τόσες δυσκολίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ράντεφ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ζήφκα για την ε, περιστατωμένη σας έκθεση. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Ε, και θα πρέπει να είναι και ε, το επίκεντρο τα παιδιά σε αυτό το θέμα. Εγώ στηρίζω αυτό που συστήνει η ε, ο κύριος Βίσκα, δηλαδή την υιοθέτηση από τη βιολική οικογένεια και επίση το, θα πρέπει να ακουστεί η γνώμη του παιδιού ως προς την υιοθέτηση. Ωστόσο θα πρέπει να σκεφτούμε και τα παιδιά, ε, τα μωρά ή τα παιδάκια 2-3 ετών που δεν μπορούν ακριβώς να εκφράσουν την επιθυμία τους και που μπορεί να απομακρυνθούν από τους ε, συγγενείς χωρίς να είναι σε θέση να αντισταθούν σε αυτή την απόφαση, να αντιτεθούν μάλλον σε αυτή την απόφαση. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και να σκεφτούμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψουμε τα παιδιά. Επίσης ε, θα πρέπει οι γονείς ε, να ε, σχετίζονται με και να συνδέονται άμεσα με τις σχετικές αποφάσεις. Η ειδική κατάρτιση δεν θα πρέπει να προσφέρεται στους δικαστές αλλά και στους κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και τους δημόσιους υπαλλήλους που ασχολούνται με θέματα υιοθεσίας στα ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προστατέψουν τα δικαιώματα του παιδιού. Όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να γίνουν με τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες. Τώρα για την αυτόματη αναγνώριση πραγματικά μου αρέσει αυτή η ιδέα του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού και θα συνέστηνα μάλιστα να είναι και πολύ γλώσσο αυτό το πιστοποιητικό ώστε το κόστος της νομιμοποίησης και το κόστος της ε, μετάφρασης να μειωθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίασή του Ωστόσο θα ήθελα να θίξω κάποια προβλήματα ε, που αφορούν τις διασυνοριακές υιοθεσίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανηλίκους, για παιδιά. Άρα το βασικό μας στόχος θα πρέπει να είναι η προστασία του παιδιού μέχρι τη στιγμή της υιοθεσίας, αλλά πιστεύω ότι και τα όσα συμβαίνουν μετά την υιοθεσία είναι εξίσου σημαντικά, γιατί κάποιες φορές έχουμε να κάνουμε με υιοθεσίες που είναι προβληματικές. Ας πούμε ένα παιδί το οποίο υιοθετείται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Το παιδί παραμένει υπό την προστασία των ε, Βρετανικών αρχών ή πρέπει να επανέλθει στη Ρουμανία κυρίως όταν οι βιολογικοί γονείς ε, επιθυμούν να ανακτήσουν το παιδί τους να πάρουν πίσω το παιδί τους. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δυστυχώς ε, συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ότι μια ρουμανική οικογένεια έχασε τα παιδιά της και τα παιδιά προτάθηκαν προς υιοθέτηση σε μια οικογένεια ομοφιλόφιλων. Αυτό επιτρέπεται ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε, εμείς διερωτηθήκαμε, μπορούμε να ξεπεράσουμε, να υπερβούμε τις αξίες της οικογένειας του παιδιού. Εγώ δεν έχω να σχολιάσω την νομική κατάσταση κάθε χώρα αλλά ωστόσο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις και σε αυτή τη διαδικασία ε, θα πρέπει να αποφύγουμε την προσβολή ε, πολιτιστικών αξιών της χώρας προέλευση, τη βιολογική οικογένεια του παιδιού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτε παιδιά τα οποία έχουν υιοθετηθεί και βρίσκονται σε τέτοιε χώρε μάλιστα που δεν είναι καν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι για μας δεν μας απασχολεί πλέον το θέμα. Πρόκειται για Ευρωπαία, ε, ε, Ευρωπαία παιδιά και μιλάω ας πούμε για την Νορβηγία και πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, να προστατεύσουμε μάλλον τα ε, συμφέροντα του παιδιού. Η Νορβηγία χαίρει σχεδόν το ιδίων, ιδίου καθεστώτος ε, που χαίρουν και οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο δεν είναι όλα ακριβώς τα ίδια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Λεμπρετό. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους ε, δύο, τις δύο εμπειρογνώμονες που μας φώτισαν. Μιλάμε για διεθνείς υιοθεσίε που είναι ένα ανθρώπινο θέμα πολύ λεπτό, πολύ ευαίσθητο και δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τις ανθρώπινες επιπτώσεις και τις απτές επιπτώσεις. Η σύμβαση του 1973 είναι καλό κείμενο, ε, κυρώθηκε από πολλά κράτη και όλα τα κράτη της Ένωσης μάλιστα. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα που υπογραμμίστηκε της αναγνώρισης της υιοθεσία που δεν είναι εξασφαλισμένα αυτή τη στιγμή. Το σημερινό κείμενο προσπαθεί να διορθώσει αυτό το θεμελιώδες πρόβλημα, όμως θα πρέπει να προσέξουμε γιατί η λύση που προτείνεται είναι να διατηρήσουμε να προσέξουμε εμείς να φτάσουμε σε ένα πολύ άκαμπτο και εξαιρετικά περιοριστικό πρόβλημα, ε, καθεστώς με συγχωρείτε. Υπάρχει ένα άρθρο 1 στο παράρτημα που επιτρέπει σε ένα κράτος να αρνηθεί την αναγνώριση της υιοθεσίας εάν αυτή η αναγνώριση είναι προφανώς αντίθετη με τη δημόσια τάξη αυτού του κράτους μέλους. Πολύ καλή διάταξη αυτή που επιτρέπει, έχω την εντύπωση, να ρυθμιστούν τα ανθρώπινα προβλήματα, σεβόμενοι ωστόσο την ιδιαιτερότητα και την κυριαρχία κάθε κράτος μέλους. Εγώ λοιπόν στη διάρκεια της συζήτησης θα με ώστε να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να σεβαστούμε την κυριαρχία κάθε κράτους μέλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάποιον άλλον να ζητά το λόγο, οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, διακεκριμένες προσκεκλημένε μα που συνέβαλαν και έτσι να κλείσουμε τη συζήτηση αυτού του θέματο και να συνεχίσουμε με το επόμενο, την επόμενη ακρόαση.